for the people who come as our yeah. guests. I know it's embarrassing. That is translation and everything. All yeah. Meine Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην κοινή συνεδρίαση της ΕΦΕΤ και ΣΕΝΤΕ. και περιμένω να δω με μεγάλη χαρά πώς θα εξελιχθεί αυτή η σημερινή ακρόαση. Ε, να μην ξεπεράσουμε τα 5-7 λεπτά ανά παρέμβαση παρακαλώ για να συζητήσουμε το θέμα των συμφωνιών του Μίνσκ. Ε, συμφωνήθηκε νομίζω ή διαπιστώθηκε στις 2 Οκτωβρίου ότι μέχρι το τέλος του έτους δεν θα μπορέσουν να συμφωνηθούν οι συμφωνίες, να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες του, του Μίνσκ. Θα δοθεί κάποια παράταση και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει κάτι τέτοιο επί των κυρώσεων. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου είναι πολύ στενά συνδεδεμένα τα θέματα. η αντίληψη είναι ότι δεν θα έρθουν σταδιακά οι κυρώσει όσο σταδιακά εφαρμόζεται η συμφωνία του Μίνσκ, αλλά όταν ολοκληρωτικά εφαρμοστούν οι συμφωνίε του Μίνσκ, τότε θα έρθουν και οι κυρώσει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι ερμηνείε αυτού του θέματο από πολιτική πλευρά. Και θα πρέπει και από τις δύο πλευρές να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Ξέρουμε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί από τη ρωσική πλευρά και η Ουκρανία δεν έχει τον έλεγχο της πρόσβασης και των συνόρων προς τη Ρωσία. Αυτό είναι αποφασιστικό σημείο, κέριο σημείο στη Συμφωνία του Μίνσκ. Δεν έχει εφαρμοστεί αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τη Συμφωνία της Δευτέρας Οκτωβρίου. Αυτά που συμφωνήσαμε για την απόσυρση ορισμένων τύπων ε, όπλων να δούμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες πρόοδοι από αυτού και τι επιπτώσεις έχουν οι εξελίξεις. Ε, μας ενδιαφέρει επίσης κατά πόσο έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία εκδημοκρατισμού ε, με την κυβέρνηση του Κιέβου και την περιφερειακή διοίκηση και αποκέντρωση να δούμε ποια είναι η πολιτική σημασία και κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για, την, για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό περιοχών όπως η Κρυμαία και να δούμε κατά πόσο η Ρωσία χρησιμοποιεί κάποια θέματα ως άλοθη. Δεν θέλουμε να δημιουργηθούν περαιτέρω περιτές εντάσεις. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι οι εξελίξεις και τι μπορούμε να κάνουμε και με την ανοικοδόμηση της χώρας. Δεν θέλουμε να δοθεί κανένα άλλο το οποίο θα είναι εις βάρος της χώρας. Πριν δώσω το λόγο η πρόεδρο της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου ε, για την ε, Ουκρανία, Μάλλον σας δίνω το λόγο για να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις, κύριε Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Έλμαρ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φωτηγά και τον κύριο Μπλοκ που οργάνωσαν από κοινού αυτή τη σημαντική ακρόαση για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες και Ευχαριστώ πολύ ε, και τον εκπρόσωπο από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι εδώ μαζί μας και από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ως πρόεδρος του του Κοινοβουλευτικού Σώματος που συναλλάσσεται με τη Φεχόφνα Ράντα μπορώ να σας πω ότι η εφαρμογή της συμφωνιών του Μίνς και είναι ένα συνεχές θέμα στο διάλογό μας, στις μερικέ διατάξει του διάλογό μας, συζητήθηκε και πριν τρεις εβδομάδες ε, στο Κίεβο με την ε, κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ε, και με τον πρόεδρο Ποροσένκο και με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και με άλλους Ουκρανούς συνομιλητές. Αυτή τη στιγμή του Μίνσκ είναι η μόνη πολιτική διαδικασία που μας ε, οδηγεί σε πλήρη και ειρηνική επανένταξη ε, με την ε, συμπερίληψη και των κατεχόμενων εδαφών στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέσκ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία και επίσης και της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΕΣΕ το έργο του νέου προσώπου, του κ. Σάιντεκ που ήρθε από τη Νέα Υόρκη ως έμπειρος αυστριακός διπλωμάτης για να βοηθήσει τη διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό, για να βοηθήσει και το έργο της κυρίας Σελαβίνη. Να πω ότι για μας είναι σημαντικό να δούμε ουσιαστικά ποιος σέβεται και ποιος δεν σέβεται τη συμφωνία. Είναι σαφές ότι η ρωσική πλευρά δεν σέβεται την ε, Συμφωνία του Μίσκου βλέπουμε τις δεσμεύσεις και βλέπουμε που υπάρχει έλλειψη πρόοδου. Επίσης, ε, παροτρύνουμε τους Ουκρανούς συναδέλφους να είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια και να αποφύγουν την κατάσταση όπου τελικά θα κατηγορήσουν αυτούς για την έλλειψη πρόοδου στην εφαρμογή της συμφωνίας. Από τη σκοπιά αυτή τους ενθαρρύνουμε να δείξουν όριμη στάση στη συνέχιση αυτής της διαδικασίας και κυρίως της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Είναι ένα κρίσιμος τομέα. Πριν κάποιους μήνες το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ε, ουσιαστικά δεν αδιακόπτουν τη εργασία τους. Είχαμε και ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ε, μπροστά από το κτίριο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακούσουμε και από τον κύριο Υπουργό τη νέα προοπτική από την Ουκρανική πλευρά. Επίσης, ανυπομονούμε να σταματήσουν οι απώλειες ζώων. Άκουσα χθε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα 32 Ουκρανοί ε, βρήκαν το θάνατο. Ε, ουσιαστικά ε, είναι λιγότερες οι απώλειες από ό,τι είδαμε από το Μίσκ αλλά και πάλι έχουμε μεγάλο ρυθμό και 8.000 ε, ζωές που έχουν χαθεί, είναι πάρα πολλές, θα πρέπει κάθε ζωή να προστατευτεί και να εφαρμοστεί κατά βαυση του πυρός πλήρως. Εμείς λοιπόν ως αντιπροσωπεία σύνδεσης με την Ουκρανία θα ενθαρρύνουμε στις, στις ε, δύο χώρες να καταβάλουν πάσα δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η λύση του προσωρινού κατεχόμενου εδάφους του Τόνπας να μην αποσυνδεθεί εντελώς από το θέμα της Κρυμαίας. Πιστεύουμε ότι η αιτία του προβλήματος είναι η ίδια. Και από τη σκοπιά αυτή δεν θα πρέπει να το παραμελήσουμε αυτό, ούτε να το παραμερίσουμε. Έτσι λοιπόν, με ισχυρή υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Προοπτική της Ουκρανίας, υποστηρίζουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και ανυπομονούμε να προβούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τους διπλωματικούς εκπροσώπους που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Αντρέη. Θα ξεκινήσουμε αμέσω με τι παρουσιάσει και θέλω να δώσω το λόγο στο Ιωάννη Ρέγκενριχτ, ε, ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία ε, πρόσωπο από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε πρόεδρε Μπροκ, αξιότιμε πρόεδρε ε, Πλένκοβιτ, αξιότιμη κυρία πρόεδρο Φωτίγκα, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση αυτή που διοργανώσατε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα προσπαθήσω να κάνω ένα σύντομο απολογισμό ο Ραφαέλ Ντελαγκάρ, άλλο συνάδελφο, ε, θα ε, περιγράψει τις προοπτικέ ε, από εδώ και πέρα και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο συγκεκριμένοι για τη διαδικασία του Μίνσκ νομίζω ότι μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει τρία πράγματα μέχρι τώρα. Πρώτον, μία στρατιωτική αποκλιμάκωση παρά της ευάλωτη εκεχηρίας. Δεύτερον, μία λειτουργική πολιτική διαδικασία και τη δημιουργία της τριμερούς ομάδας επαφής στο Μίνσκ που κάθε εβδομάδα σχεδόν συναντώνται οι ομάδες εργασίας ε, για πολιτική, ανθρωπιστικά ζητήματα και θέματα όπλων και ασφάλειας, τρεις ομάδες εργασίας. Ε, υπό την αιγίδα των κρατών της Νορμανδίας όπως ονομάζονται και εκφράζονται πολλά συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα προγράμματα για την οικονομία, για την ανοικοδόμηση της χώρας και παρότι είναι δύσκολες ε, οι περιστάσεις, ε, σημειώνονται πρόοδοι. Υπάρχει η προσωπική δέσμευση της καγκελαρίου Μέρκελ και του Προέδρου Ολάντ και με τους Υπουργούς Εξωτερικών Μάιε και Φαμπίρις και με όλες αυτές τις διαδικασίες ε, προσπάθησαν να προωθήσουν τις συμφωνίες ε, του Μίνσκ. Ε, ήταν μεγάλη στρατιωτική αποκλιμάκωση. Κατάφεραν δηλαδή να αποτρέψουν μια κλιμάκωση ε, στρατιωτική και παρά τα πολλά άλλα προβλήματα, παρά τη Συρία, παρά την τρομοκρατία, παραμένουν προσιλωμένοι στο θέμα της Ουκρανίας γιατί γνωρίζουν ότι η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας δεν έχει εκλείψει, θα παραμείνει και γι' αυτό παραμένει και το θέμα στο επίκεντρο. Χρειάζεται να παραμείνουμε προσιλωμένοι στους στόχους της συμφωνίας του Μίνσκ και στην υλοποίηση των συμφωνιών αυτών. Είναι δύσκολη η διαδικασία της ε, εκεχηρίας μέσω ε, των εξελισσομένων ε, διαδικασιών βλέπουμε πόσο πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν στη διαδικασία, πόσο ευάλωτη είναι αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε την πλήρη υλοποίηση ε, των συμφωνιών, απόρριση των βαρέων ε, όπλων, απόρριση των ελαφρών όπλων, συνεχιζόμενη εκεχηρία και τοπικές εκλογές στον Ταμπάς και αυτό θα μας οδηγήσει σε ε, μια βελτίωση της κατάστασης. Τα βασικά ε, στάδια σε αυτή τη διαδικασία είναι ε, μια επαληθευμένη εκεχηρία που θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2016 να έχει ολοκληρωθεί να μπορέσει, όπως είπε ο πρόεδρος Μπρόκ, να έχει έλεγχο των συνόρων η Ουκρανία και να μην παρεμβαίνουν παράτυποι παραστατιωτικοί σχηματισμοί. Παραμένουν οι συμφωνίες του Μίνσκ στο προσκήνιο και θα ήθελα εν συντομία να μιλήσω για τη συμφωνία της απόσυρσης των όπλων και των ανθρωπιστικών ζητημάτων και τις προοπτικές στην πολιτική διαδικασία με την ε, κεχηρία της πρώτης ε, ενάτου ε, είχαμε κάτι το οποίο λειτουργήσε επί δύο μήνες σχετικά καλά όμως από τα τέλη Οκτωβρίου άρχισαν κάποιες, άρχισε μια αύξηση των παραβιάσεων της ε, κεχηρίας, ιδίω στην περιοχή του Ντανιέτσκ, φαίνεται ότι αυξάνεται αυτή η τάση και καθ' όλη τη διάρκεια ε, του Νοεμβρίου είχαμε περισσότερες παραβιάσεις της εκεχηρίας από ό,τι τον Οκτώβριο. Αυτό οφείλεται στο ότι οι συμφωνίες για την απόσυρση των όπλων και από τις δύο πλευρές, ιδίω από την πλευρά των αποχιστικών, ε, κινημάτων αλλά και από των Ουκρανών, δεν εφαρμόζονται ε, κατά τρόπο θα έπρεπε μέχρι τις 11-12 Νοεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί. Ο ΑΣΕ δεν ε, έχει ε, καταφέρει να διαπιστώσει πλήρη υλοποίηση αυτών των συμφωνιών, διότι πολλά όπλα δεν έχουν δηλωθεί και ε, είναι πίσω από την διαχωριστική γραμμή και διακινούνται ελεύθερα, θα μπορούσε να πει κανείς τα, ε, ο βαρύς οπλισμός με διαμέτρημα πάνω από 20 χιλιοστά ε, ε, είναι αντικείμενο της συμφωνίας επίσης. Ο ΑΣΕ προσπαθεί να επιτύχει επιτυχία και δηλώθηκαν μέχρι χθε χίλια τέτοια οπλικά συστήματα και θα πρέπει να δηλωθούν και να δηλωθεί και ο τόπο απόσυρση για να μπορεί να γίνει η επαλήθευση τη απόσυρση. Χρειάζεται λοιπόν μια πλήρη συμφωνία για την απόσυρση των ελαφρών και των βαρέων όπλων. Αν δεν γίνει αυτό δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα. Επόμενη προτεραιότητα είναι η άρση των ναρκοπεδίων και εδώ υπάρχουν ε, μεγάλες δυσκολίες. Πριν από δύο εβδομάδες ε, ε, είχαν γίνει κάποιες συμφωνίες για τις προτεραιότητες που θα δοθούν και για τους τομείς προτεραιότητας για την αποναρκοθέτηση και η ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΣΕ είναι ιδιαίτερα διστακτική ως προς τα αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος του έτους δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και αυτό έχει σχέση ε, και με τα ανθρωπιστικά προγράμματα και με τις διαχωριστικές γραμμές. Τώρα για το ανθρωπιστικό πρόγραμμα θα ήθελα να πω κάτι. Ο πρέσβης Τόνι ε, Φρίστ είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας, ε, είναι από την Ελβετία συντονιστής του προγράμματος και δουλεύει με την ομάδα εργασίας Οικονομία μαζί με τον Φίσερ που είναι και ο Γερμανός συντονιστής. Έχουμε κοινά προγράμματα για την ανθρωπιστική δράση. Καταγράφονται οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Υπάρχουν οι επιτόπου γιατροί χωρίς σύνορα. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επίσης είναι ενεργή επιτόπου. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα σημεία διέλευσης, να ανοίξουν περισσότερα ε, σημεία διέλευσης και να μπορούν να περάσουν και πέρα από, ε, από τη διαχωριστική γραμμή. Το Μάιο και τον Ιούνιο δεν είχαμε καμία προθυμία για συνομιλίες, αλλά από το καλοκαίρι και μετά υπάρχει βελτίωση και υπάρχει συνεργασία είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν οικονομικές πρωτοβουλίες στην Ουκρανία και να μην αφήσουν τους Ρώσους ε, να μπλοκάρουν τις περιοχές ε, ε, όπου υπάρχουν τα αποσχιστικά κινήματα. Ένα ζήτημα είναι η πληρωμή συντάξεων από την Ουκρανία, από τα ασφαλιστικά ταμεία της Ουκρανίας, αυτή είναι μια δέσμευση που είχε αναλάβει να υποστηρίξει η Γαλλία και η Γερμανία στις συμφωνίες ε, του Μίνσκ και έχουν δημιουργηθεί κέντρα λογιστικής ε, με τερματικά τραπεζών και η κρατική τράπεζα, η USAID, ε, ε, δίνει πρόσβαση στους συνταξιούχους για να μπορεί η Ουκρανία να καταβάλει τις συντάξεις. Ε, επίσης, μια γερμανική αποστολή προσπαθεί να επαναφέρει το πόσιμο είδος στην περιοχή του Λουγκάνσκ και του Ντανιέσκ και επισκευάζει τις, τα κατεσταμένα δίκτυα ίδρευσης Επίσης τις κατεστραμμένες ε, σιδηροτροχές ε, και τις ε, κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Προσπαθούμε λοιπόν με τα έργα ανασυγκρότησης να δημιουργήσουμε μια θετική κατάσταση και για τις δύο πλευρές. Είναι λοιπόν θετικές οι προοπτικές, υπάρχει συνεργασία, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες προκλήσεις τώρα στο τέλος του έτους και στην επόμενη χρονιά. Και όπως είπε και ο πρόεδρος Βρόκ, αυτό έχει άμεση επιπτώσεις επί των κυρώσεων. Ολοκληρωτικά θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί η συμφωνία του ΜΙΝΚ για να μπορούν να αρθούν οι κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις ε, που ισχύουν μέχρι τις 31 ε, ε, πρώτου. Για την Κρυμαία υπάρχουν κίνδυνοι για την ηλεκτροδότηση λόγω της καταστροφής του δικτύου έχει υποχρέωση, υπάρχει υποχρέωση παράδοσης για την Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους και ελπίζουμε ότι θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση για να μπορεί να υπάρχει παροχή μέχρι το τέλος του έτους και να μην έχει και καμία πρόφαση η Ρωσία εναντί της Ουκρανίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, κύριε Πρόεδρε των σχέσεων με την Ουκρανία, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη δημόσια αυτή διαβούλευση. Οι συνάδελφοι μου, ο Γιώργος Ράγκιο Μπρέχτ και εγώ, έχουμε έρθει για να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση εφαρμογή των συμφωνιών του ΜΙΚ και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να υπογραμμίσω την εξαιρετική συνεργασία μας με τη Γερμανία σε κάθε επίπεδο μεταξύ της ε, Καγκελαρίου και του Προέδρου μας μέχρι το χαμηλό επίπεδο το δικό μας UKNS. Ποια είναι, ποιες είναι οι προπτικές. Προτεραιότητά μας φυσικά παραμένει η ενίσχυση της κατάστασης της ε, ασφάλειας επιτόπου και η εφαρμογή των διαφόρων πλευρών των συμφωνιών του ΜΙΣΚ που ε, θέλουν να ενισχύσουν την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση ασφάλειας που είναι οι δύο πλευρές του δύο νομίσματος και βεβαίως προσπαθούν να επαναφέρουν την απαραίτητη ε, εμπιστοσύνη στις πολιτικές συζητήσεις και βεβαίως χρειάζεται μια πολιτική διαδικασία για να δρεωθεί η κατάσταση πυρός, πράγμα που δυστυχώς έχει, η έλλειψή της μάλλον έχει οδηγήσει σε πολλές παραβιάσεις από τις αρχές Νοεμβρίου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καθόρισαν μια αλληλουχία της ε, υλοποίησης των ε, συμφωνιών του Μίνσκ. Αυτό πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στη διάρκεια ε, συνάντησης κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 2 Οκτωβρίου του 2015 και βεβαίως ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στην όλη διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από την αρχή της, των συμφωνιών Μίνσκ. Αυτή η αλληλουχία προβλέπει τα εξή. Καταρχήν, την ε, καταγγελία των αυτονομιστών στις εκλογές που μονομερώς διακήρυξαν και βεβαίως την ε, ε, επιβεβαίωση των, μιας συγκεκριμένης ημερομηνία. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Δεύτερον, η προώθηση μια, ενός νέου νόμου, ειδικού νόμου για τις εκλογές σε περιοχές που, τις οποίες αφορούμε και η οποία θα εφαρμοστεί από το ραντάρ, αλλά αυτό θα επανέλθω στις, ε, στην, στο πολιτικό σκέλος η πραγματοποίηση εκλογών 90 μέρες μετά την ψήφιση αυτού του νόμου, κατόπιν η παρουσίαση υποψηφίων, κατόπιν η θέση ενισχύ της αμνηστίας μετά τις εκλογές και πάρα πολύ σημαντικό κατόπιν η θέση ενισχύ του νόμου για το ειδικό καθεστώς διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, σε περιοχές του Ντονιές και του Λουγκάνς, την περιοχή της των εκλογών προψωρινά καταρχήν και κατόπιν θέση ενισχύ οριστικά την ημέρα όπου η, η οργανισμός ο ΑΣΕ θα αποφασίσει ότι είναι αδιαμφισβήτητη η εκλογική διαδικασία. Η ομάδα εργασίας για τα πολιτικά θέματα που συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, Τρίτη και ε, Τετάρτη στο Μίνσκ συνήθως με τα εμπλεκόμενα μέρη, Ουκρανούς, Ρώσους και τους αυτονομιστές, τις δύο οντότητες και ε, που είναι υπό τον συντονιστή του ΟΑΣΕ, αυτή η ομάδα εργασία συνεχίζει για να ε, εντοπίσει κρίσιμες παρα, παραμέτρους για τις τοπικές εκλογές στις δύο αυτές ζώνες. Οι παράμετρες αυτοί είναι γνωστές και έχουν αναγνωριστεί και την έχουν, τις έχουν επαναλάβει οι Υπουργοί Εξωτερικών στο Βερολίνο στην Υπουργική Συνάντηση που έγινε μετά την ε, συνάντηση κορφής του Παρισιού στις 2 Οκτωβρίου, δηλαδή στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε αυτό στο Βερολίνο. Και, και μετά το, τη συνάντηση αυτή ο Γερμανός Υπουργός υπενθύμησε τις παραμέτρους και, τους, και τις ρυθμίσεις. Πρώτον, η σεβασμό στα δικαιώματα των ε, εκτοπισμένων. Δεύτερον, συμμετοχή πολιτικών κομμάτων. Τρίτον, ελεύθερη πρόσβαση των μέσων ενημέρωση. Τέταρτον, η, ε, Παρατηρητέ στις εκλογές και τέλος ε, αποτέλεσμα των εκλογών. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις, ε, στα πρότυπα του ΟΑΣΕ όπως προβλέπει ευθύς εξ αρχή το πακέτο μέτρων για την υλοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ. Εκ παραλίλου ε, και βεβαίως πάντοτε σύμφωνα με τις συμφωνίες του Μίνσκ οι Ουκρανικές αρχές έχουν αναλάβει να ξεκινήσουν μια ε, αναθεώρηση του συντάγματος, συνταγματική διαδικασία που αφορά την αποκέντρωση. Ε, και στο πακέτο Μίνσκ γίνεται αναφορά ε, στην ιδιαιτερότητα των ζωνών Μίνσκ, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Και βεβαίως αναφέρεται, το κείμενο αυτό το συντάσσει μια ε, Ουκρανική Επιτροπή. Θα σας μιλήσει ο Ουκρανός συνάδελφος και θα περάσει από δεύτερη ανάγνωση στη Ράντα με, με ειδική πλειοψηφία. Εκεί βρισκόμαστε όσον αφορά τη διαδικασία στην Ουκρανία. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε ε, τους αυτονομιστές οι οποίοι συμμετέχουν πραγματικά επικοδομητικά στις ε, διαδικασίες της ε, πολιτικής ομάδας της συνεργασίας για να φτάσουμε στις τοπικές εκλογές σε, συντονισμό με το Κίεβο και σύμφωνα με, τις, με την νομοθεσία της Ουκρανίας και με βάση τα επίπεδα του ΟΑΣΕ σύμφωνα με το, τις αποφάσεις του Μίνσκ στις 12 του περασμένου Φεβρουαρίου. Και βεβαίως περιμένουμε η Μόσχα να εξασκεί την επιρροή της στους ε, αυτονομιστές όπως έγινε κατά την, δήλωση, την, την κοινή δήλωση για την υποστήριξη του πακέτου Μίνσκ. Η διαδικασία αυτή θα, θα ευοδοθεί εάν ε, πλαισιώνεται και από ένα πακέτο. Και εδώ σας υπενθυμίζω την δέσμευση όλων των πλευρών και ιδιαίτερως της Γερμανίας και της Γερμανίας με πάρα πολλές συναντήσεις, πολλές ε, τηλεφωνικές επαφές που έγιναν ε, από την αρχή της διαδικασίας αυτής. Έκτοτε από τότε που ξεκίνησαν όλα αυτά, η δέσμευση ε, στο πλαίσιο της Νορμανδίας από όλες τις πλευρές είναι σαφής. Οι επόμενες ε, επαφές δεν έχουν ξεκινήσει στη φάση αυτή. Είμαστε στο, ε, έγινε η Υπουργική στο Βερολίνο στις 6 Νοεμβρίου και από εκεί και πέρα τις επόμενες ημέρες, πριν τα Χριστούγεννα εν πάση περιπτώσει, θα γίνει μια άλλη επαφή ε, υψηλού επίπεδου στο πλαίσιο Νορμανδίας. Τώρα η διαδικασία Νορμανδίας έχει κάπως, όπως ξέρετε υπήρχε μια αρχική προθεσμία 31 Δεκεμβρίου 2015, de facto έχει παραταθεί για λίγους μήνες αυτή. Έχει έχει, αυτό έχει αποφασίσει από κοινού ο πρόεδρος Δημοκρατίας, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Ποροσέγκο και ο πρόεδρος Πούτιν στο, στο Παρίσι στις 2 Οκτωβρίου. Και μετά από αυτή την αλληλουχία που σας περιέγραψα συμφώνησαν για μια προθεσμία 90 ημερών για την οργάνωση των εκλογών από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος στην Ουκρανία, δηλαδή από τις 2 Οκτωβρίου έχει κάπως καθυστερήσει πέρα, δηλαδή ξεπερνά την προθεσμία της 31 η Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, αποφασίσουν για την ανανέωση των οικονομικών ε, ε, κυρώσεων ε, που λήγουν στις 31 Ιανουαρίου 2016 και αυτά είναι τα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου. Έτσι πρέπει λοιπόν στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό να γίνει μια συζήτηση για την ανανέωση αυτών των κυρώσεων που σας περιέγραψα. Ε, πέρα από αυτή την προθεσμία και έχοντας γνώση όλες τις όλων των δυσκολιών που πρέπει να ξεπεραστούν ε, μας ενδιαφέρει η διαδικασία συνέχισης οργάνωση τοπικών εκλογών στις ζώνες των αυτονομιστών θέλει να ενισχύσει την ασφάλεια και να συνεχίσει η πορεία απομάκρυνσης των ναρκών όπως ακούσατε. Ε, τώρα, το πέρασμα, η ψήφιση του νόμου του ειδικού νόμου για τις περιοχές και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι, έχει δυσκολίες και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Τέλος, ε, ε, χρειάζεται και μια επένδυση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΕ για την πολιτική διαδικασία. Πριν κλείσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω τι έχει κάνει η Ουκρανία το ε, την πορεία που οδήγησε και τις δυσκολίες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί όλα αυτά προχωρούν παράλληλα με μια άνευ προηγουμένου διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία, κυρίως στον τομέα της οικονομίας ε, και, τις, το και, τις, τα δημοσιονομικά. Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλοί νόμοι από την Άνοιξη, ε, ε, νόμοι που αφορούν την ε, μείωση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και, της, και δημοσιονομική νόμη. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν, αποτελούν θετική πορεία στα πλαίσια της... Ε, ε, έναρξης της ισχύω της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο και ευχαριστώ και τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας ε, για την δέσμευσή τους μέσω της οποίας ε, βοηθήσατε να σταματήσει η στρατιωτική διαδικασία και ξεκίνησε μια πολιτική διαδικασία που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να φτάσουμε σε μια ειρηνική λύση. Και από τις δύο αυτές παρεμβάσεις είδαμε πως ε, υπάρχει σαφής δέσμευση για την υλοποίηση των συμφωνιών ε, του Μίνσκ. Είναι ξεκάθαρη η θέση και δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Και τώρα δίνουμε το λόγο στον Όλεξη Μακέλεφ, πολιτικό διευθυντή από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, εξωτήμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα πολύ να είναι ο άνθρωπος που θα σας ε, ανέφερε ότι εφαρμόζεται η Συμφωνία του Μίνσκ και ότι έχει επιστρέψει η ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα επιτόπου είναι εντελώς διαφορετική. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, όπως ε, σωστά είπε ο κ. Σπανκοβίτς, Ανησυχούμε τώρα με τις ε, προκλήσεις της στρατιωτικής της Ρωσίας. Η Ρωσία υποστηρίζει παράνομες ένοπλες ομάδες ε, και έχουν δική τάση. Από το 29 Αυγούστου έχουμε πάνω από 1.100 βομβαρδισμούς των θεσεών μας, πυροβολισμούς κατά των θεσεών μας και επίσης υπήρξαν και 14 ενόπλες προκλήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε ε, 37 στρατιωτών στην Ουκρανία και πολλούς τραυματίες και έχουμε τουλάχιστον 18 αμάχους ε, που κατέληξαν. Και παρά τις υποσχέσεις της Ρωσίας στο Παρίσι σε υψηλότερο επίπεδο και στο Βερολίνο σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών οι μαχητές είτε πλήρως είτε μερικώς περιορίζουν την πρόσβαση της ειδική αποστολής παρατήρησης του ΑΣΕ στα εδάφη τα οποία τώρα είναι από τον έλεγχο των Ρώσων και των αντιπροσώπων τους ε, ε, ουσιαστικά ο ρόλος της αποστολής ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός προκειμένου να παρατηρήσει πως είναι κατάσταση επιτόπου και να εγγυηθεί την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας απόσυρσης. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα, η έλλειψη ασφάλειας ε, θέτει αρνητικό ιστορικό την στιγμή που τέσσερι υπουργοί συμφώνησαν στο Βερολίνο ότι η πολιτική ομάδα εργασία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τέσσερα κυρία στοιχεία σε ό,τι αφορά τι τοπικέ εκλογέ στον Ντόνμπα. Γιατί οι τοπικέ εκλογέ είναι το τελικό στάδιο τη όλη πολιτική διαδικασία. Εμεί θέλουμε να εκλέγονται οι άνθρωποι και να εκπροσωπούν την περιφέρεια εκεί και δεν θέλουμε ανθρώπους να διορίζονται από τη Μόσχα για να κυβερνούν. Τα κυρία στοιχεία αυτών των συνομιλιών για τις εκλογές είναι το να επιστρέψουν εσωτερικά εκτοπισμένοι. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένους στην Ουκρανία και κάθε ένας από αυτούς των 1,5 εκατομμύριο έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλέξουν τους τοπικούς τους εκπροσώπους. Δεύτερον, αυτό αφορά το σχηματισμό εκλογικών επιτροπών. Επίσης, πρόσβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάθε ε, Ουκρανός, ε, Ρώσος, ε, εκπρόσωπος των μέσων και από άλλες χώρες έχει δικαίωμα να μεταβεί στην περιοχή. Επίσης, η συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων της Ουκρανίας στις εκλογές είναι απαραίτητο. Όλοι στην Ουκρανία έχουν δικαίωμα και του εκλέγει και του εκλέγεσθε στις τοπικές εκλογές. Και φυσικά το να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλείας και για τους πολιτικούς και για τους ψηφοφόρους και για τους διεθνείς παρατηρητές. Υποθέτω ότι όχι μόνο οι παρατηρητές του ΑΣΕ αλλά και οι εκπρόσωποι του οίκου αυτού θα κληθούν σε αποστολή παρατήρηση των εκλογών. Έτσι λοιπόν θέλουμε ασφάλεια για όλους. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση. Δυστυχώ οι μαχητέ συνεχίζουν να μπλοκάρουν τι δραστηριότητε των διεθνών οργανισμών επιτόπου. Το ανέφερε αυτό και αναφέρθηκε στους γιατρούς χωρίς σύνορα που δεν τους επιτρέπεται να εργαστούν εκεί. Επίσης, οι αυτονομιστές συνεχίζουν να γνωρούν το ότι συμφωνήθηκε στο Μίνσκ για την απελευθέρωση όλων των αχμαλώτων αμέσως. Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς, εξακολουθούμε να έχουμε δέκα κρονούς αχμαλώτους που κρατούνται στη Ρωσία ως πολιτικοί αχμάλωτοι και θα πρέπει να απελευθερωθούν. Οι ε, ε, αντιπρόσωποι της Ρωσίας ε, θυμός της Ρωσίας στον Τόνμπα συνεχίζουν να παραβιάσουν τη διαδικασία της εφαρμογής του Μίνσκ. Πρέπει να ασκήσουμε ενοποιημένη πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία και οι αυτονομιστές θα σταματήσουν τις προκλήσεις και θα διασφαλίσουν πλήρη κατάπαυση του πυρός. Δεν θέλω να διαβάζω πλέον σε εκθέσεις για θύματα από το μέτωπο. Επίσης, ε, να σεβαστούν το θέμα της απόσυξης του βαρέως αλλά και του ολιφρού οπλισμού και να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος του SMM, δηλαδή της αποστολής του ΑΣΕ. Να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στην όλη επικράτεια και να δοθεί πρόσβαση στον έλεγχο των συνόρων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Πάνω από 400 χιλιόμετρα των συνόρων αυτών δεν είναι υποέλεγχο αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ένα μεγάλο παράθυμα για να εισαχθεί από εκεί νέος επιλεσμός, νέοι μαχητές και φυσικά προσωπικό του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας. Βάσει της λογικής των συμφωνιών του ΜΙΣΚ να ακολουθηθεί η λογική αυτή και να ακυρωθεί το αποτέλεσμα των των εκλογών που έγιναν στον Τόνμπας το 2014. Επίσης να συμφωνήσουν να γίνουν τοπικέ εκλογές σύμφωνα με την Ουκρανική νομοθεσία στο εγγύ μέλος και να απεμπλοκαριστούν οι δραστηριότητες όλων των διεθνών οργανισμών. Να σας πω και δύο λόγια για τις δραστηριότητες της αποστολής του ΕΦΕ. Αυτή η ομάδα των παρατηρητών που νομίζω ότι τώρα πλέον από 700 άτομα, κάνει πολύ καλή δουλειά στο να παρακολουθεί την κατάσταση. Βάζουν τα δυνατά τους. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσουν την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να υποστηρίξετε εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ιδέα της εφαρμογής ε, το να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αποστολή που θα επιτηρεί για την εφαρμογή των συμφωνιών του ΜΙΣ και θα προετοιμάσει μια πολιτική λύση για το όσα έχουν συμφωνηθεί στο Μίνσκ. Αυτή η αποστολή θα χρειαζόταν επίσης και για την οργάνωση και την διενέργηση των τοπικών εκλογών σε τελικό στάδιο. Για να συνοψίσω. Η Ουκρανία παραμένει δεσμευμένη στην πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Εμείς θέλουμε να επανέλθει η ειρήνη και πιστεύω ότι όλοι σε αυτό τον νοίκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμφωνούν με αυτή την πεποίθηση. διαδικασία της διαβούλευσης στο Μίνσκ, οι δραστηριότητες ε, του, της ομάδας της Νορμανδίας ε, είναι ζωτικά στοιχεία για την εξέβριση λύσης και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας, Γερμανίας και Γαλλίας στην Ορμανδία, στο πλαίσιο της ομάδας συνομευτής. Στο τέλος της παρουσίασης αυτής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Τώρα τι κάνουμε στην Ουκρανία αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας και πιστεύουμε ότι υποστήριξη στον αγώνα μας από το Βερολίνο, από το Παρίσι αλλά και από τις Βρυξέλλες και από κάθε μεμονωμένη πρωτεύουσα είναι σημαντική. Θα θέλαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός, τα κράτη-μέλη και ο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν όχι μόνο το Ουκρανικό κράτος αλλά και τους Ουκρανούς στον αγώνα μας για ελευθερία, στον αγώνα μας για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αξιών, προκειμένου να γίνουμε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό κράτος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίγκαν, διευθυντή τη ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ και τα μέλη τη Επιτροπή ε, για τη συνεργασία μα ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα εξ αρχή αρχής να δηλώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τις συμφωνίες του Μίνσκ Χαιρετίζουμε τις σημαντικέ προσπάθειες οι οποίες γίνονται από δύο κράτη-μέλη με μεγάλες επενδύσεις πολιτικού κεφαλαίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει συνολικά τον σεβασμό της για την κυριαρχία της Ουκρανίας και αυτό αποτυπώνεται και στην υποστήριξη προς τις ε, συμφωνίες με των οποίων δεσμεύεται η Ουκρανία. Ε, ε, διακυβεύεται η κυριαρχία και η ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Παράλληλα, τίθεται σε κίνδυνο και η σύνδεση με την Ουκρανία, διότι δεν θα θέλαμε να παρατείνεται μια κατάσταση σύραξης σε μια συνδεδεμένη χώρα εταίρο, την Ουκρανία δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, άλλη μία μετασοβιετική συνεχή σύραξη. Ο στόχος μας ε, είναι να βρεθεί ένας τρόπος να ρυθμιστεί η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία μέσα στο συνταγματικό και νομικό πλαίσιο της Ουκρανίας και θα πρέπει να αφιερώσουμε ε, μεγάλη ενέργεια στο να επιλύσουμε και το θέμα της προσάρτησης της Κρυμαίας. στην Υπουργική Διάσκεψη του ΟΣΕ στο Βελγράδι ε, σήμερα, γιατί η Αντιπρόεδρος ε, Μογκερίνη αυτή τη στιγμή μιλάει εκεί, κάνει την παρέμβαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει πολλές ε, διπλωματικές και πολιτικές επαφές με τον κύριο Λαμπρόφ και με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Παρασέγκο με πανότατους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η υποστήριξη δεν είναι μόνο διπλωματική. Είναι και πολύ συγκεκριμένη, υποστηρίζει διαδικασίες και πέραν της διαδικασίας στο πλαίσιο της Νορμανδίας και είναι και πρακτική υποστήριξη. Στις συνομιλίες καταφέρουμε να επιτύχουμε μια δεύτερη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και την ασφάλεια στον ε, ενεργειακό εφοδιασμό τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά το χειμώνα και συνεχίζονται και οι συνομιλίες ε, της CFTA όπου ελπίζουμε ότι θα έχουμε πρακτικές, πρακτικά αποτελέσματα πριν από τα τέλη του έτους, αν και είναι δύσκολο πολλές φορές να συμφιλιώσουμε θέσεις που μοιάζουν ασυμφιλίωτες. Η πρακτική υποστήριξη συνίσταται στην σημαντική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ειδική αποστολή παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Τα δύο τρίτα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε δώσει 25 εκατομμύρια από κονδύλια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Επίσης δίνουμε σημαντική βοήθεια για καταρχήν ανθρωπιστική βοήθεια. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι πάνω από το ίμιση της ε, βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία στο πλαίσιο της ε, σύγκρουσης αυτής ε, πηγαίνει σε περιφέρειες που δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Δεν περιορίζεται λοιπόν η ανθρωπιστική βοήθεια μόνο σε αυτό το τμήμα της Ουκρανίας αλλά πηγαίνει και σε άλλα τμήματα της Ουκρανίας. Δίνουμε τώρα ένα τεράστιο πρόγραμμα υποστήριξη για τη διαδικασία αποκέντρωση στην Ουκρανία και θα παράσχουμε υποστήριξη επίση για τη διακυβέρνηση και για την αποκατάσταση της ειρήνης ε, μέσω του προγράμματος ανάπτυξης ε, των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή του Ντανιέσκη και του Λουχάνσκα 97 και 10 εκατομμύρια επιπλέον και δίνουμε σημαντική βοήθεια και για την άρση των ναρκοπαιδείων. Θα αποτελέσει μίζωνα προτεραιότητα στο μέλλον, ένα από τα απαραίτητα βήματα, αφού, όπως είπε ο κύριος Ρέγκενμπρεχτ, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο. Η δυσκολία στην υλοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ Εκτός από την ε, αρχική δυσκολία που είναι έλλειψη πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση των συμφωνιών είναι ότι υπάρχουν και διαφορετικές ε, πλευρές, ε, οικονομική, πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική. Θα έπρεπε να είναι αλληλοσυμπληρούμενες πτυχές, αλλά πολύ συχνά είναι πτυχές οι οποίες μπλοκάρουν η μία την άλλη. Αν δεν υπάρχει πρόοδος σε ένα τομέα, δεν μπορεί να προχωρήσει η πρόοδος και σε άλλο τομέα. Και θέλω να τονίσω την ε, ανάγκη ε, να βρεθεί κάποια λύση για τις ε, τοπικές εκλογές. Αυτό θα αποδεσμεύσει και πολλά περαιτέρω βήματα. Τονίσαμε την σημασία της επιτυχίας της συνάντησης του Παρισιού και την ε, Υπουργική Συνάντηση, αλλά όπως είπαν οι συνάδελφοι υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν αυτές τις τοπικές εκλογές υπό διεθνή ε, επιτήρηση συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και με παρακολούθηση από τα μέσα ενημέρωση. Υπάρχουν δύσκολα θέματα σε σχέση με το ρόλο τη Κεντρικής εκλογική Επιτροπής και των τοπικών εκλογικών επιτροπών. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Πλένκοβιτ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έχουν γίνει ε, στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεση. Η Ράντα θα πρέπει να ψηφίσει τον, την τροποποίηση του συντάγματος για την αποκέντρωση ε, και τον νόμο για τις τοπικές εκλογές καθώς και ένα ειδικό νόμο για τις ε, ε, διατάξεις αυτοδιοίκησης ορισμένων περιοχών του Ντανιέτσκ και του Λουχάνσκ. με την ε, έναρξη μια σειρά συνομιλιών ε, για την απόσυρση ξένων ε, στρατευμάτων και για τη δημιουργία θεσμών ελέγχου των συνόρων από την Ουκρανία θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Είναι μια δέσμη μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Όπως ήδη είπαν ο Γάλλος και ο Γερμανός συνάδελφος, είναι ε, ε, σαφή τα σημεία που έχουν οριστεί από τους αρχηγούς κατών και κυβερνήσεων δηλαδή πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως οι συμφωνίες του Μίνσκ για να μπορέσουμε να λάβουμε θετικές αποφάσεις για μια πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων Αυτά είναι τα ορόσημα που έχουν τεθεί αν η υλοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ χρειαστεί περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί τι περισσότερο χρόνο και για τα, ε, τις υπόλοιπες αποφάσεις εκ μέρου μα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες ε, που έχουμε κοντά μας ε, και θα σας δώσουμε το λόγο στη συνέχεια για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η βασική στάση της Ρωσίας ενάντια της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει. Είναι ρεβιζιονιστική και οπορτουνιστική. Εκμεταλλεύεται την ευκαιρία η, οποία, η οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται με πολιτικά κίνητρα. Είναι θετικό το ότι υπάρχουν οι συμφωνίες του Μίνσκ και ότι προσπαθούμε να επιτύχουμε σωστά αποτελέσματα. Είχα πάει στην Ουκρανία το φθινόπωρο και η συζήτηση που γινόταν είναι τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν έχουν υλοποιηθεί οι συμφωνίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει προσιλωμένη η Ουκρανία στο να υλοποιηθούν οι συμφωνίες μέσα στην επόμενη χρονιά. Πότε προβλέπεται η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική τροποποίηση στο, Φερχόβνα Ράντα. Πιστεύω ότι το πολιτικό μήνυμα πρέπει να είναι ότι ίσως για την παρούσα φάση κάτι μπορεί να αναβληθεί, αλλά ε, με τη ρωσική πολιτική του Πούτιν δεν ξέρω τι πρόοδο μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό ίσως πρέπει να ενθαρρύνουμε τους Ουκρανούς ε, να προχωρήσουν. Όσον αφορά τις εκλογές, πώς θα διεξαχθούν τεχνικά όταν πρέπει να συμμετάσχουν στις εκλογές και οι εκτοπισμένοι με λεωφορεία θα μεταφερθούν για να ψηφίσουν αυτοί που είναι εκτοπιστέντες ε, με επιστολική ψήφο, πώς θα γίνει. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν πολλές ακόμη πτυχές ε, που οδηγούν σε συγκρούσεις. Ε, ο εφοδιασμός σε φυσικό αέριο, διάβασα ότι διακόπη από τη Ρωσία, οι αεροπορικές μεταφορές θα έχει αποκατασταθεί η, αεροπορική, η εναέρια κυκλοφορία, απαγορεύεται η υπερπτήση. αν θέτουν περαιτέρω απαιτήσει από τη ρωσική πλευρά, ποια θα είναι η εξέλιξη. Αυτές είναι οι βασικέ ερωτήσει. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να αφιερώσουμε όλο το χρόνο για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις του κ. Γκάλα. Δίνω το λόγο όμως και σε άλλο ομιλητή, ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Μάλλον ρώτησε, είδε τι ερωτήσει μου ε, από και ο προηγούμενο ομιλητή και έκανε όλες τι ερωτήσει που θέλω να κάνω κι εγώ. Ποιε θα είναι οι προτεραιότητε που θα θέσετε μέσα στην επόμενη χρονιά, τι ρόλο παίζει ο ΑΣΕ, πώς βλέπετε την κατάσταση και τι πρωτοβουλίες θα υπάρξουν από τη γερμανική πλευρά που θα βοηθήσουν στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Thank you. Next, Mr. Tan. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έχει πάρα πολλές κρίσεις να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς δεν έχουμε επικεντρωθεί όσο θα πρέπει στην ε, ε, επιθετική πολιτική της Ρωσίας στην Δυτική Ουκρανία και την Κρυμαία δεδομένου ότι μας έχει απασχολήσει περισσότερο το θέμα της και τώρα υπάρχει το, ε, το ε, δημοψήφισμα. Όμως όπως είπε και ο, ο Ουκρανός διπλωμάτης δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συμφωνίες του Μίνσκ χωρίς να έχουν λυθεί τα θέματα με τη Ρωσία στα σύνορα και ε, οι, οι, οι ρωσικές κυρώσεις στην Τουρκία ε, μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους πώς θα επηρεάσουν την, την κατάσταση όσον αφορά τη βοήθεια που προσφέρει η Τουρκία στους διοκόμενους τάταρους αδερφούς τους. Ε, υπάρχει υπάρχουν ε, πολύ σοβαρά θέματα που αποτελούν σχεδόν ε, πυρηνική απειλή. Τώρα, Όσον αφορά την Κρυμαία ε, και την κατάσταση εκεί θα υπάρξει αύξηση ε, της επιθετικότητας της Ρωσίας, η δυνατότητα να αυξήσει η Ρωσία την επιθετικότητα μέσω τη Μαριούπολης και βεβαίως ποιες είναι οι πιθανότητες επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Ρωσία και προσπαθεί τώρα η Ρωσία να ενισχύσει τη θέση της στη Βιέννη λόγω της εμπλοκής της στη Συρία. Επίσης υπάρχει καμία διάθεση για να υπάρξει η ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την παρακολούθηση και πώς ε, θα εφαρμοστεί η DCFTA η οποία σύντομα θα αρχίσει να τίθεται ενισχύει. Πώς θα εφαρμοστεί στην Κρυμαία. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ απαιτητική, αλλά έχουμε ακριβώς 40 λεπτά για αυτή τη συζήτηση ε, που πρέπει, στην οποία πρέπει να απαντήσουν και οι ομιλητές. Λοιπόν, δεν θέλω να σας, ε, να σας πιέσω, αλλά σας παρακαλώ προσπαθήστε να είστε πάρα πολύ σύντομοι, κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συνήθως σύντομος, ναι. Εκτιμώ το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση Θέλω όμως να επισημάνω ότι λείπει ένα πολύ σημαντικό ε, κομμάτι ε, που λείπει ε, και που αφορά πολύ σημαντικό, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο την, για την υλοποίηση του Μίνσκ, Μίνσκ 1, 2, 3 και δεν ξέρουμε πόσα, που ξέρουμε ποιο είναι αυτός ο υπεύθυνο εταίρος ο οποίος έκανε την προσάρτηση. Ξέ, οι διατάξει υλοποίηση του Μίνσκ, των συμφωνιών Μίνσκ, έχουν άμεση σχέση με τι κυρώσει. Είναι πάρα πολύ λογικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες της Δύση έκαναν ε, κυρώσει έκαναν κυρώσεις, υπέβαλαν κυρώσεις κατά το επιτιθέμενου. Η διαδικασία του Μίνσκ περιλαμβάνει και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Μην ξεχνάμε ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας, ε, δηλαδή μια χώρα έχει ε, διαμελιστεί. Μιλάμε λοιπόν για κυρώσει, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Charles Τένοξ στην ερώτησή του. Όταν δούμε τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι συμφωνίες του Μίνσκ, δηλαδή ε, μεθοριακή έλεγχη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπάρξει υλοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ. Οπότε ε, ε, απευθύνω την ερώτησή μου σε προσώπους των κρατών μελών. Βλέπετε ότι υπάρχει ε, δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη με αναφορά στις αποστολές CSDP οι οποίες ενδεχομένως θα αναπτυχθούν γιατί είναι χρήσιμες. Ευχαριστώ κύριε Σαπχάουζα. Κυρία Πρόεδρε, με καταρχήν που ε, η, το πλαίσιο της Νορμανδίας περιορίζεται. Ξεχάσαμε κάποιον, τη Ρωσία. Δεν είναι το τι κάνει συνήθως, τι κάνουν συνήθως ο κύριος Ολάντ, ε, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Ποροσέγκο, ξεχνούν τη Ρωσία. Εγώ έχω, το έχω συνηθίσει αυτό. Έχω συνηθίσει να μην είναι αντικειμενικές οι επιτροπές μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ένωσης γιατί ο κ. Βίγκαν είχε ε, μια πολύ ισορροπημένη παρουσίαση. Δεν έχω συνηθίσει να ακούσω ισορροπημένες παρουσιάσεις. Ε, συνήθως ακούω ότι όλο το βάρος πέφτει στη ρωσική πλευρά και ένας είναι ο υπεύθυνος η Ρωσία θέλω να πω στον, στον Γάλλο, όχι συνάδελφο αλλά συμπατριώτη μου, ότι όταν λέει ότι θα ήταν απαραίτητο να υποστηρίξει η Ρουσία με όλη της τη δύναμη την ειρήνη, θα μην ξεχνάμε τις Ηνωμένε Πολιτείε, να μην ξεχνάμε το πραξικόπημα που είχε προετοιμαστεί νωρίτερα. Μην ξεχνήσουμε την κυρία Νούλαντ, η οποία επιβάλλει την θέλησή της στην Ευρώπη χρειάζονται δύο συνομιλητές και πρέπει πραγματικά να μην χρησιμοποιείται ε, η σύγκρουση στην ε, Ουκρανία. Χθε ακούσαμε τον κύριο Μακόβεν, έναν πολύ διάσημο αναλυτή της CIA, τον οποίο γνωρίζω και ο οποίος μας το υπενθύμησε αυτό. Ελπίζω να το θυμόσαστε και να έχετε κατά νου τις πληροφορίες που μας έδωσε. Θα ήθελα να πω στον ε, εκπρόσωπο της Ουκρανίας ότι εγώ έχω συμμετάσχει στις εκλογές ως παρατηρητής, όπως θα το γνωρίζετε, στο Ντόνετσκ και δεν είδα άτομα τα οποία έχει ορίσει η Μόσχα. Είδα ανθρώπους που κινητοποιούνται και εκλεγμένους. Είδα όμως εκεί που τώρα γίνονται εκλογές όλους τους εκπροσώπους της κυβέρνησής σας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους απορρίφθηκαν. Αυτή είναι η, η, αλήθεια. Οι ελεύθερες εκλογές είναι τέλειο. Αλλά σας ρωτάω, γιατί δεν περιμένατε κι εσείς τόσο πολύ να περάσει αυτός ο νόμος για την αποκέντρωση που θα επιτρέπει ώστε να γίνουν αυτές οι ελεύθερες εκλογές. Γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επιμένω ότι από εξ αρχής. Ναι, ναι, θα ολοκληρώσω, ναι. Θέλω να, να πω ότι ευθύ εξ αρχή πίστεψα στι συμφωνίε του Μίνσκ, συνεχίζω να τι πιστεύω και είμαι βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία ειρήνη και ότι σε αυτήν πρέπει να συνεισφέρουμε έχοντα ένα ε, ε, μια ακριβή εικόνα της, των ε, ευθυνών κάθε πλευράς. Ευχαριστώ κύριε Σκόπιν. <clears throat> Άκουσα τον, ε, μάλλον συγγνώμη έχασα ένα μέρος της ομιλίας του κυρίου Ντελαγκάρτ. Μου λείπουν κάποιες, ε, κάποια στοιχεία, κάποιες πληροφορίες. Όταν μιλάτε για ειδικούς ε, για διευθετήσεις, αυτές οι ειδικές διευθετήσεις ισχύουν μόνο για το Λουγκάνσκ και τον Ντονέσκ ή σε όλες τις περιφέρειες της Ουκρανίας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν έχουμε ξεχωριστή μεταχείριση για αυτές τις δύο περιοχές είναι σαν να τις διαφοροποιούμε από την υπόλοιπη Ουκρανία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από πολιτική σκοπιά. Ευχαριστώ. Κύριο Σκέλαμ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπε ο συνάδελφος ε, Στρίβιτς διδίδασε ε, το κύριο μένυμα Όμως ε, ουσιαστικά ακούσαμε ότι υπάρχουν 400 χιλιόμετρα ανεξέλεγκτων συνόρων. Και άλλα στοιχεία των συμφωνιών του Μίνσκ ε, ουσιαστικά δεν θα υλοποιηθούν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα κύρια σημεία του Μίνσκ. Όμως αυτό είναι πακέτο και χωρίς να ελέγχουμε τα ανατολικά σύνορα νομίζω δεν υπάρχει και τίποτα άλλο που μπορεί να γίνει. Και μια ακόμη ιδέα. Η Ρωσία ενδιαφέρεται πολύ για να έχει ένα συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτου ε, στη Μέση Ανατολή. Μπορούμε να στείλουμε στους Ρώσους το μήνυμα ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο συνασπισμό αν δεν υπάρχει πληρή εφαρμογή των συμφωνίων του Μίνσκ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλα. Συμφωνώ μαζί σας. Επόμενος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ. Κρίμα που βγήκε ο κύριος Σαφχάουσερ. Γιατί μίλησε για το ότι λείπουν εδώ κάποια κράτη από τη συζήτηση. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι λείπουν και πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάμε και για όμορες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η δική μου χώρα συνορεύει και με τις δύο αυτές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίσει και τα περιφερειακά συμφέροντα των κρατών στον τομέα της ε, ασφάλειας, ε, γιατί αυτό ε, δεχόμαστε μεγάλες απειλές από αυτή τη σύραξη. Έχω δύο ερωτήσει προς τους ομιλητέ. Καταρχήν, Πώ βλέπετε την κατάσταση στην Πεσσινατολή γιατί υπάρχει και ένα θέμα εδώ δικαιώματος της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών. Αυτό ισχύει για την Ουκρανία φυσικά. Τελικά χάσαμε τη στιγμή που έπρεπε να δράσουμε και τώρα αυτή η αντίδραση θα είναι πολύ πιο δύσκολη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε έτσι ώστε οι απειλές εξ Ανατολής ε, να συνιστήσουν απειλή κατά κατάσταση ασφάλειας ε, των ανατολικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω και μια ρητορική ερώτηση. Δεν πιστεύετε ότι η κατασκευή του North Stream 2 γίνεται ουσιαστικά κομικοτραγική και είναι και κομικοτραγικές και κυρώσεις που εφαρμόζεται. Αν μπορεί η Ρωσία ε, με τη Δυτική Ευρώπη να περασπίσει τα ζωτικά της συμφέροντα, Πού είναι οι πολιτικές και οικονομικές πιέσεις για τις οποίες μιλάμε. Και η τρίτη μου ερώτηση για τον εκπρόσωπο της Ουκρανίας θα ήθελα να σας πω ότι σας υποστηρίζουμε πλήρως και για το να συσταθεί μια αποστολή επιτήρησης που θα επιτρέψει να ελέγξει την εφαρμογή της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς προφέρονται τα ονόματά σας. Έτσι λοιπόν με συγχωρείτε για ενδεχόμενα λάθη. Κύριε Στάκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά το είπα το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές ε, και θεωρώ πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Ήδη έχουν πει πολλά οι συνάδελφοι πριν από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η αξιολόγηση από την πλευρά των Ευρωπαίων συναδέλφων σχετικά με τις κυρώσεις. Ε, Ενδεχομένω υπάρχουν κάποιες προκλήσεις. Και δεύτερον θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την ε, υλοποίηση του DCFTA, της Ειρικής και Ισβάθος Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Μιλήσαμε για ε, τις συνέπειες της Συμφωνίας του ΜΙΣΚ και τις συνέπειες του DCFTA και της Συμφωνίας Σύνδεσης δεν ήταν πολύ επικοδομητικές, πολύ αποδοτικές τέλο πάντων οι συζητήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ποια είναι η αξιολόγησή σας, οι εμπορικές συμφωνίες θα υλοποιηθούν όπως θα όφυλαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να μην υπάρξουν περιττές καθυστερήσεις οι περιπλοκές. Καταλαβαίνουμε βέβαια τη, σημασία των συμφωνιών του Μίνσκ. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Οι συμφωνίε του Μίνσκ είναι η μόνη μας ελπίδα να δούμε κάποια λύση στην κρίση αυτή. παρακολουθούμε τις εργασίες των συναδέλφων στη Ράντα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ήδη έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Όμως παραβιάζονται συνεχώς οι συμφωνίες του Μίνσκ. 11 Φεβρουαρίου συνήθισαν οι συμφωνίες του Μίνσκ, ήμουν παρόν τότε και είδα ήδη από την πρώτη μέρα υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις και έκτοτε υπάρχει μεν μία αποκλιμάκωση, αλλά ήδη χτες μια δήλωση του Γιάννου Σότεμπεργκ, Γενικού Γραμματέα του ε, ΝΑΤΟ, ε, επισήμανε ακριβώς τα προβλήματα αυτά. Είπε ότι υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος να ξαναρχίσουν οι βιοπραγίες στην Ανατολική Ουκρανία παρόλε τι προσπάθειε για την υλοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ. Υπάρχει κίνδυνο επανέναρξη λοιπόν των σειράξεων. Τώρα, για τι εκλογέ. Η Ράντα έχει παράξει νομοθετικό έργο. Υπάρχει εσωτερική διαδικασία στο Κίεβο, αλλά χρειάζεται και υποστήριξη επιτόπου. Διαφορετικά θα πάνε χαμένες οι προσπάθειες. Δεν θέλω να φαίνομαι απεσιόδοξος, αλλά ε, και σε μια ακρόαση για στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιλούσαμε για την αποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Λουχάνσκο όπου υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξοι. Ε, υπάρχει κάποιο ψήγμα αισιοδοξία, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές. Ακούσαμε ε, ε, στην ε, γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες το γερουσιστή που έλεγε ότι δεν θα τηρηθούν οι συμφωνίες μέχρι τέλους του έτους αλλά αυτό το έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει και πολλές φορές έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αν η Ρωσία συνεχίσει να υποστηρίζει θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους αυτονομιστές μπορούμε να είμαστε εμείς αισιόδοξοι ποιος πιστεύει ότι η Ουκρανία θα ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων της. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι αυτό θα είναι ένα σημείο κλειδί για να κλείσει η Συμφωνία Μίνσκ 2 και ποια είναι η νέα προθεσμία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τη γνώμη σας για όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Βάτλαντ. Ε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ στα Ολλανδικά. Αφού παρακολούθησα ολόκληρη τη συζήτηση Ακούσαμε για την ανθρωπιστική κρίση, την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης κλπ. Αυτά που είπε ο κύριος Μάκιεφ λένε ότι η Ρωσία συνεχίζει τις παραβιάσεις. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε περισσότερο πίεση στη Ρωσία. Πώς θα το καταφέρουμε. Ήδη έχει ασκηθεί αρκετή πίεση. Αν αυξηθεί, θεωρώ ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να ε, πλαισιώσουμε τη συμφωνία του Μίνσκα, αλλά δεν βλέπουμε ποιο τρόπο. Υπάρχει η, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι, θέλουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις αποστολές, αλλά αυτό Πώς πιστεύετε ότι θα γίνει, ε, δηλαδή πιστεύετε ότι θα το επιτρέψει αυτό η Ρωσία, θα το διευκολύνει, θα, μπορέσει να υπάρξει συγκεκριμένη ανάθεση εντολή στην αποστολή η οποία να θα, τις οποίες οι εργασίες θα ευοδοθούν παρακολουθώντας τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν Πιστεύω ότι θα πρέπει ίσως να κάτσουμε και να συζητήσουμε ότι εμείς επηρεαζόμαστε από τις κυρώσεις πολύ από την πόλη μου πολλά προϊόντα εξάγονται στη Ρωσία, πληττόμαστε λοιπόν και θα θέλουμε, ε, θέλει ο πληθυσμός να μάθει τι συμβαίνει γιατί είναι θύματα ενός πολέμου με τον οποίο δεν έχουν καμία σχέση. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στον πόλεμο στη Συρία, τις επιθέσεις στο Παρίσι. Έχω την εντύπωση ότι έχει υπάρξει πλέον ε, ε υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν την ισορροπία. Η συζήτηση για τη Συρία θα πρέπει να μας βοηθήσει να ε, ζητήσουμε από τη Ρωσία να αλλάξει στάση απέναντι στο Μίνσκ και την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, ε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη επειδή δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τη συζήτηση στα Ισπανικά. Μπορείτε όμως να μιλήσετε Ισπανικά και θα μεταφραστεί η ομιλία σας. Έχουμε παθητικά Ισπανικά στο γλωσσικό σύμβο της Συνεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φωτήρα. Θα ήθελα να κάνω διάφορες ερωτήσεις. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ενημέρωση από την πλευρά της Επιτροπής και το λέω ειλικρινώς, είμαι 48 χρόνια ως δικηγόρος εργάζομαι και πάντοτε πριν ε, να υπάρξει αποτέλεσμα, ακούμε τα μέρη. Φυσικά ένα από τα μέρη εδώ είναι η Ουκρανία. Έλα, άλλο μέρος ε, στο Μίνσκ, καλά και στην Ορμανδία είναι η Ρωσία. Εγώ θέλω να ζητήσω η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να έχει τη λογική της ουδετερότητας ότι όταν μιλάμε ε, για τα μέρη, τα μέρη να είναι μέρη και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και η Ρωσία μπορεί να μας έδινε κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εγώ θεωρώ ότι τα σύνορα της ε, Ουκρανίας έχουν καθοριστεί στη Βουδαπέστη και στο Ελσίνκι. Είναι ξεκάθαρη η θέση μου λοιπόν, αλλά νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να ακούσουμε για να καταλάβουμε και δεν το κάνουμε. Αυτή η Επιτροπή μόνιμα είναι απομακρυσμένη από το ένα από τα μέρη της σύραξης. Δεύτερον, αν θέλουμε ε, να δούμε τι θα γίνει με την καβολή της συντάξεων από την νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας στο Λουγκάς και στο Ντονές και με τον ίδιο τρόπο να δούμε τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα που θα πρέπει να δοθεί στους Ουκρανούς πολίτες. Δεύτερον, ε, φυσικά δεν τηρείται η κατάπαυση του πυρός, απλώς θέλουμε να, πρέπει να δούμε αν γίνεται αυτό μόνο από την πλευρά των αυτονομιστών ή και από τις δύο πλευρές. Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν όσοι χρηματοδοτούνται από ολιγάρχες αυτές οι ομάδες έχουν διαλυθεί και, ε, ή στην Ουκρανία έχουν ενταχθεί στις κανονικές ενόπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και δεν είναι υπό τη δίκαιωση ολιγαρχών. Ανησυχώ επίσης ε, για στην έκθεση της ε, Transparency International σε σχέση με την Ουκρανία. Λέει ότι υπάρχει γενικευμένη διαφθορά. Εγώ ως δικηγόρος ε, ξέρω ότι άλλο είναι ο νόμος και άλλο η πραγματικότητα. Εμένα με ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας νόμος που να επιτρέπει και να προωθεί την ε, διαφθορά. Όμως θα ήθελα να μου πείτε σε ποια, ποια είναι η κατάσταση. Γιατί η έκθεση της Transparency International μιλούσε για κάτι πολύ ανησυχητικό. Ότι ο πληθυσμός στην Ουκρανία αντιλαμβάνεται ως κάτι φυσικό τη δωροδοκία και τη διαφθορά και μάλιστα θεωρούσε ότι δεν εκπροσωπείται από τους πολιτικούς. Και η εκλογική διαδικασία είναι παθολογική. Ουσιαστικά βλέπουμε ε, ότι τι συμβαίνει στην, στην περιοχή. Έχουμε διαφορετική κατάσταση στη Δύση και στις ανατολικές περιοχές. Στις ε, προεδρικές εκλογές μόνο το 59% των πολιτών στην Ουκρανία ψήφισαν, ενώ ότι το 1999 είχαμε το 65% του πληθυσμού στις κοινοβουλευτικές, το 62% ε, ενώ υπήρχε μείωση και στις σημερινές τοπικές εκλογές το 46% και στο δεύτερο γύρο το 34% συμμετείχε. Έτσι λοιπόν κοινωνιολογικά η κατάσταση μου φαίνεται πάρα πολύ ανησυχητική. Απομακρύνονται οι πολίτες από τους πολιτικούς τους εκπροσώπους. Thank you, for... Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Ουσιαστικά εδώ μιλώντας εξ ονόματος των εκλογιών μου. Θα ήθελα να πω όσα υπόθηκαν από τον κύριο Μάρα Από τον Πίτερ, Αστραβίτσιους και από όλους τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που προέρχονται από την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Ακούγοντας τις παρεμβάσεις σας, Ουσιαστικά κατάλαβα ότι είμαστε μαζί με το Ουκρανικό έθνος. Φυσικά όμως ε, σκεφτόμαστε και τη μοίρα των δικών μας χωρών, των δικών μας εθνών. Και συνειδητοποιούμε ότι αυτή η κατάσταση στην Ουκρανία απειλεί την ασφάλεια και στην ευρύτερη περιοχή μας και ξέρουμε ποιος φταίει. ξέρουμε ποιο είναι το μέρος που φταίει. Έφυγαν οι δύο συνάδελφοι, ο κύριος Αφχάζος και ο Νάρα, όμως ήθελα να τους πω ότι η Ρωσία έχει πολλές δυνατότητες να προωθήσει τη θέση της, ενώ εμείς, ακόμη και αν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πολύ λίγες δυνατότητες να απαντήσουμε Χαίρομαι πολύ που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει κάποιες δράσεις και που μπορέσαμε να ακούσουμε και το Γάλλο, το Γερμανό διπλωμάτι και φυσικά χαιρετίζω εδώ και τον κύριο Διευθυνταή και τον κύριο Μακέφ. Είμαστε μαζί σας. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Βίγκαν, θα ήθελα να πω ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δεν είναι κάτι που τίθεται σε αμφισβήτηση. Έχει παραβιαστεί. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και τώρα, πάλι υπό το ρόλο μου ως πρόεδρος, θα δώσω το λόγο καταρχήν στους δύο διπλωμάτες που εκπροσωπούν τη Γερμανία και τη Γαλλία και τα Υπουργεία Εξωτερικών. Παρακαλώ κύριε Ρέγκερμπερτ και κύριε Ντελαγκάρτ. Έχετε καταρχήν το λόγο και κατόπιν ο κύριος Μακίεφ και ο κύριος Βίγκαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σαφώς υπάρχουν ε, προκλήσεις ενώπιον μας και πολλές ερωτήσεις ε, σήμερα. Θα προσπαθήσω να επιλέξω τις ερωτήσεις που αφήνονται περισσότερο ε, στη Γερμανία. Και ζητώ συγγνώμη αν κάποιες από τις ερωτήσεις σας δεν τις απαντήσω ή δεν τις απαντήσω πλήρως. Έχω σημειώσει λοιπόν κάποια σημεία στα οποία θα απαντήσω. Πρώτον, για τη διαδικασία του Μίνσκ και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Θα ήθελα να πω το εξή. Ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση, ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση αν αφήναμε μόνη τη την Ουκρανία και αν επιτρέπαμε την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Θα καταλήγαμε σε άλλη μια παγωμένη σύραξη στην Ευρώπη, όπως η Υπερδνηστερία, η ε, Νότια Οσετία, η ε, Αφχαζία, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ε, με προβλήματα για την ακαιρεότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Αυτά πρέπει να είναι και ο στόχος για μας. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη συμφωνία αυτή χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας και γι' αυτό Περνώ στην επόμενη ερώτηση για το ρόλο του ΑΣΕ και της Γερμανίας. Στο Βελιγράδι σήμερα θα είναι θέμα προτεραιότητας ε, ε, αυτό στις συζητήσεις ε, του ΑΣΕ και στην Ουκρανία παίζει κεντρικό ρόλο και στο πλαίσιο της τριμερούς ομάδας επαφής εξασφαλίζει το συντονισμό και μέχρι τώρα ήταν πολλές οι επιτυχίες της ε, ειδική Επιτροπής Επιτήρησης. Παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες ε, να αποκατασταθεί ο διάλογος και προσπαθούμε να ε, ε, συμμετάσχει και η Ρωσία. Η Ρωσία είναι ένας από τους εταίρους στη διαδικασία της Νορμανδίας και θα πρέπει ε, ξεκάθαρα να πούμε τι πιστεύουμε για το ρόλο που έχει παίξει η Ρωσία σε την ε, διένεξη. Το βλέπει διαφορετικά η Ρωσία, αλλά εμείς ε, πιστεύουμε ότι η Ρωσία είναι ένας από τους εμπλεκομένους της διένεξης αυτής. Δεύτερο ερώτημα, τα σύνορα. Ο στόχος των συμφωνιών του Μίνσκ είναι το να έχει η Ουκρανία πλήρη έλεγχο ε, των ε, συνόρων που έχουν μήκος πάνω από 400, πάνω από 400 χιλιόμετρα. Ε, και ο Ρεξέη Μακίεφ ε, ανέφερε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να έχουμε την διαδικασία των εκλογών πρώτα και την αποκατάσταση της κυριαρχίας της Ουκρανίας στα σύνορά της στη συνέχεια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Προς το παρόν έχουμε την ειδική αποστολή παρακολούθηση που πρέπει να την ενισχύσουμε για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές κατά μήκος των διεθνών συνόρων και θα δούμε πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και να ενταθεί. Τρίτο σημείο, η Κρυμαία. Παραμένει προτεραιότητα και οι κυρώσει θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η παράνομη προσάρτηση της Ρωσίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά παράλληλα γνωρίζοντας και θέματα της παραβίας των δικαιωμάτων των Τατάρων της Τουρκίας θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ε, για την ενίσχυση του διαλόγου και για την αποκατάσταση ε, των ε, κατεστραμμένων δικτύων και, της, και για την επάνωδο της φυσιολογικής ζωής στην περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε εφαρμογή των συμφωνιών από τις αρχές του έτους και θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ε, καμία δυνατότητα στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει ε, την DCFTA ως πρόφαση. Από τις αρχές του επομένου έτους θα αρχίσει ε, να ισχύει η συμφωνία για να μην ε, παρέχει κανένα άλλο στη Ρωσία. Θα παραμείνουμε προσυλλομένοι στο θέμα της Ουκρανίας, στην σταθεροποίηση και στις μεταρρυθμίσεις. Η διαφθορά είναι σαφώς ένα πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα των ολιγαρχών στην ε, Ουκρανία. Κύριε Μακίεφ, γνωρίζετε τα προβλήματα εσείς που δουλεύετε επί τόπου και χρειαζόμαστε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων που θα είναι πιστική και αποτελεσματική για να μπορούμε να βελτιώσουμε τα ελλείμματα που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά δεν θα αφήσω καθόλου χρόνο στους συναδέλφους να απαντήσουν. Ευχαριστώ, στη Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα πολυάριθμα ερωτήματα. Θα τα πάρω με τη σειρά. Από τον κύριο Καλέμπριο για την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία. Τους νόμους, την συνταγματική αναθεώρηση, αυτά τα αφήνω στον Ουκρανό συνάδελφο. Αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω είναι ο σημαντικός για σας ρόλο, επειδή είσαστε ευρωβουλευτές, με τις επαφές σας και τη συνεργασία σας από τη Ράντα. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω. Επίσης ρωτήσατε για το φυσικό αέριο και αυτό αφήνω τον Ουκρανό συνάδελφο. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κρίση στον τομέα αυτό και πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός Ουκρανίας είπε ότι σκοπίμως η Ουκρανία δεν αγόρασε ρωσικό αέριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω. Για την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών πολλές ερωτήσεις ετέθηκαν σχετικά. Πρόκειται να τεθεί εν ε, ισχύ την 1η η του 2016 και γίνονται τριμερείς διαπραγματεύσεις. Πρόσφατα ε, ε, έγινε πριν από δύο μέρες ε, μια συνάντηση. Φυσικά πλησιάζουμε την ημερομηνία θέσεως ενισχύως. Ενισχύει. Τώρα, κύριο κύριος Ε, κυρώσεις της Ρωσίας κατά της Τουρκίας που αφορούν τη Συρία και τη Μέση Ανατολή είναι θέματα που επανέρχονται συχνά. Επ' αυτών των δύο θεμάτων θέλω να επενθυμίσω ότι για τη Γαλλία η προτεραιότητα ε, που αποδίδει στην ε, αντιδρομοκρατική δράση δεν επηρεάζει καθόλου την προσπάθεια να βρεθεί μια λύση στην πολιτική κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτά είπε και την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος ε, πρόεδρος όταν συναντήθηκε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Κατόπιν, ο κύριος Οστροβίτσιους και φοβάμαι ότι μπερδεύω τα ονόματά σας, μην ξεχνάμε την προσάρτηση της Κρυμαίας. Βεβαίως δεν ξεχνάμε την Κρυμαία παρότι δεν βρίσκεται στο πλαίσιο που έχει ανατεθεί στο Μίνσκ. Η Γαλλία ε, έχει καταδικάσει την παράνομη προσάρτηση Κρυμαίας. Ε, είχατε και ένα δεύτερο ερώτημα για τα ευρωπαϊκά μέσα για την υλοποίηση των συμφωνιών είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Θέλω να σας πω ότι ήδη υπάρχουν κάποια μέσα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, η αποστολή παρατηρητών του ΟΑΣΕ, επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή σε κάποια σημεία της Μεθορίου Ρωσίας-Ουκρανίας, υπάρχει το θέμα ε, των εκλογών και της ε, των παρατηρητών του ΟΣΕ θεωρώ ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα και να, συνεργα... δουλέψουμε κυρίως για την αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ που κάνει εξαιρετική δουλειά στο πεδίο όμως πρέπει να εργάζεται ε, συνεχώς ο κύριος Σαφάουζερ, συμπατριώτης μου που μίλησε για πραξικόπημα. Εγώ μιλούμε, εμείς μιλούμε περισσότερο για επανάσταση. Αυτό είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η ίδια η ε, Ουκρανική κυβέρνηση και η Ρωσία. Μιλήσατε για την Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν τον ξεχνάμε. Συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία καθημερινά στο πλαίσιο της Νορμανδίας, των τεσσάρων της Νορμανδίας. Ε, μιλούμε και με τους ε, Αμερικανούς εταίρους και έχουμε και άλλους εταίρους στην Ευρώπη και βεβαίως τα, διεθνή θεσμικά όργανα. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε από κοινού μια συνεργασία να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Συνεχίζω. Ο κύριος Γιούρεκ από την Πολωνία για τη Μέση Ανατολή. Σας απήντησα σχετικά με τα δύο αυτά ζητήματα που είναι εντελώ χωριστά. Αναφερθήκατε στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είπα. Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και εμείς και ο ΑΣΕ. Η κυρία Σάπκα, η οποία νομίζω δεν βρίσκεται εδώ, για τις κυρώσεις για να επενθυμίσουμε πού βρισκόμαστε ε, θα ξεκινήσει μια συζήτηση για τις κυρώσεις γιατί λίγουν στις 31 Δεκεμβρίου θα γίνει μια συζήτηση επί τη βάση ενός εγγράφου Μία ερώτηση για την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών απήντησα πάλι, πρόκειται να τεθεί ισχύ την 1η Πρώτου 2016. Ερώτηση του κυρίου Μίκερ ε, για τη βία και άλλες σχετικές ερωτήσεις. Πραγματικά η κατάσταση δεν είναι ρόδινη. Υπάρχουν δυσκολίες. Πραγματικά όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Βλέπουμε τη διαδικασία της ασφάλειας και τη διαδικασία σε πολιτικό επίπεδο είναι συνδεδεμένες. Υπάρχει μια φάση Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου φέτος όπου διαπιστώσαμε σαφή βελτίωση της κατάστασης στο πεδίο με μείωση του αριθμού παραβιάσεων της κατάστασης του πυρός και έγιναν και προόδοι στο πολιτικό πεδίο με την απελευθέρωση αυτής της ε, αλληλουχίας στο Παρίσι της 2 Οκτωβρίου και το ειδικό καθεστώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά προχωρούν μαζί και εδώ και λίγες εβδομάδες από τις αρχές Νοεμβρίου και πάλι υπάρξει, έχει υπάρξει υποβάθμιση της ε, υπο, ε, επιδείνωσης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας. Βλέπουμε ότι και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος στο πολιτικό σκέλος. Αυτά ο, έχει φύγει ο Ισπανός βουλευτής, αλλά μίλησε η Τροσία, νομίζω ότι απήντησα. Τα σύνορα, οι μεθόριος βεβαίως αναφέρθηκαν, υπάρχει έλεγχος του μεθορίου στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μίνσκ είναι ο τελικός μας στόχος. Α, ο, ο, ο βουλευτής από την Ισπανία ρώτησε για τη διαφθορά. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση Ουκρανίας έχει ξεκινήσει μεταρρυθμίσει, θα ξεκινήσει και άλλε και για την ε, δικαιοσύνη, την αστυνομία, τη δημόσια διοίκηση, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίω δεν αποδίδουν άμεσα, αλλά αυτό που έχει σημασία για μα είναι να στηρίξουμε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Προσπάθησα να απαντήσω στι περισσότερε ερωτήσει και τώρα δίνω το λόγο στον Ουκρανό συνάδελφο. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχετε χρόνο κύριε Διευθυντά. Έχουμε 25 ερωτήσει και 3 λεπτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα κάνω τη δήλωσή μου κραπτός. Περαιτούμε τη δηλώσή μου. Μάλιστα, θα απαντήσω εν συντομία σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ε, στεναρή υποστηρίξη της ιδέας αυτής, ότι αν δεν ε, υπάρξει κατάσταση του ελέγχου στα σύνορα δεν μπορεί να υπάρχει τελική λύση της σύραξης. Δυστυχώς όλα τα μέσα και τα στοιχεία που προτείνουμε στη Ρωσική Ομοσπονδία για να ξαναξεκινήσει σταθερά επανέλεγχο των συνόρων, τα αρνήθηκε η Ρωσία. Καταρχήν είχαμε τον SMM ε, που μπορούσε να φτάσει κατευθείαν στα σύνορα και να αξιολογήσει την κατάσταση, αλλά μπλοκαρίστηκε την ε, αποστολή παρατηρητών του ΕΣΕ που βρίσκεται τώρα σε δύο σημεία διέλευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος. Αυτή τη στιγμή και πάλι αρνήθηκε η Ρωσία να παρατείνει την εντολή αυτής της αποστολής παρατηρητών να την επεκτείνει για το συνολικό έλεγχο των συνόρων με το μήνυμα δεν θέλουμε να ελέγχεται σύνορα δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το παράθυρο του λαθρεμπορίου όπλων στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της τελικής λύσης και σας ευχαριστώ που το υποστηρίζετε. Κύριε Γκάλερ, ε, είχατε κάνει μια ερώτηση για το αν ισχύουν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Παραμένουν σε ισχύ και δεσμευόμαστε στην εφαρμογή τους μέχρι την εξέβριση της τελικής λύσης. Όλα τα μέρη της Νορμανδίας ε, το ήθελαν αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν να εργαζόμαστε από αυτού, αλλά όπως ξέρετε χρειάζονται και τα δύο μέρη να συμμετάσχουν. Θα πρέπει και η Ρωσία να είναι επικοδομητική, να είναι στο τραπέζι και αν χρειαστεί θα πρέπει να παροτρινθεί για να συμπεριφερθεί ανάλογα και να συνεισφέρει στην εξέβρεση τελικής λύσης και να μην καταπατήσει τις συμφωνίες του Μίνσκ. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεισφέρει στο να παρατηρεί πλέον τη Ρωσία. Οι κυρώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο και είναι σημαντικό να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευμένη στο να βοηθήσει την Ουκρανία να εφαρμόσει κοινωνικέ και οικονομικέ μεταρρυθμίσει στη χώρα. Και πάλι την άκληση στου Ευρωπαίους εταίρους να σκεφτούν την επέκταση τη παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου για να βοηθήσουν την Ουκρανία στο να αντιμετωπίσει δύσκολε καταστάσει κατά μήκο των συνόρων με τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά το μήκο τη γραμμή επαφή Για τις μεταρρυθμίσεις τώρα στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση αυτή και η Φερστιφέχοφνα Ράντα, εμείς δεν χρησιμοποιούμε την επίθεση της Ρωσίας ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι. Είναι πρόκληση αυτή για μας, αλλά είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό. Αυτή είναι η μοίρα μας και με τη δική σας βοήθεια θα μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα. Και να φέρουμε ένα νέο αίμα σε όσους πιστεύουν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες μπορούν να διαδοθούν και σε άλλες χώρες. Οι άνθρωποι που βγήκαν στο δρόμο το 2014 πέθαναν όχι επειδή υπήρξε πραξικόπημα αλλά επειδή κρατούσαν ευρωπαϊκές σημαίες και ονειρεύονταν για τη χώρα μας ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Dr. Ξέρω ότι μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε εσά. Και σας παρακαλώ να περιορίσετε την παρέμβασή σας στο δυνατόν περισσότερο. Και εγώ εξάλλου το ίδιο θα κάνω. Απλώς θα ευχαριστήσω τους διπλωμάτες, το Γάλλο και Γερμανό πρέσβη που ήρθαν σήμερα εδώ. Το θεωρώ ε, κίνηση ευγένεια εκ μέρου του. Δεν είναι σύνηθε να έρχονται διπλωμάτε εδώ και κατανοώ ε, την ε, ευγενική διπλωματική χειρονομία. Στο πλαίσιο της εθνικής διπλωματίας είναι πιο εύκολο γιατί υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ είναι περισσότερο διπλωματικές οι σχέσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις παρατηρήσεις που, για τις παρατηρήσεις που κάνατε. Κύριε Βίγαντ, σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν και ένα λεπτό θα το εκτιμούσαμε. αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει το χρόνο ομιλίας για αυτά τα θέματα και εμείς ε, θα υποβάλουμε γραπτό στα σχόλιά μας. Θα σας διευκολύνω, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί οι προλαλήσαντες έχουν δώσει πολλές απαντήσεις. Πρώτον, η CFTA

Δεύτερον, αν άλλα θέματα θα ε, υπερκαλύψουν το θέμα της Ουκρανίας ε, υπάρχει μεγάλη κρίση στη Συρία ναι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση έχουμε εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης Τουρκίας. Ε, ε, εμφανίζεται ο κίνδυνος της τρομοκρατίας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση κρατών και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα πολλές προκλήσεις. Αυτό δεν, ε, δεν είναι πρωτοφανές. Είχαμε στο παρελθόν θέματα με την Ελλάδα και θέματα με το ευρώ και είχαμε και θέματα με την Ουκρανία. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματα ανάλογα με τις απαιτήσει του κάθε θέματος. Τρίτον, η αναθεώρηση των κυρώσεων. Οι συνάδελφοι το έθεσαν. Το Συμβούλιο θα προχωρήσει σε αποφάσεις ε, σύντομα. Αφού έχουν διατυπώσει τις, ε, τις ανάγκες του αρχή κρατών και κυβερνήσεων. Τώρα έχουμε μια αποστολή στο Κίεβο, η οποία τώρα μετά την ε, στρατηγική επανεξέταση θα μπορέσει να λειτουργήσει διαφορετικά. Υπάρχει ε, και λειτουργική στήριξη, όχι μόνο στρατηγικές συμβουλές. Προτείνω όμως να πούμε ότι αυτός είναι, αυτή είναι μια αποστολή για την αναθεώρηση του πολιτικού ε, κλίματος. Δεν πρέπει να ζητήσουν τα κράτη-μέλη να στείλουν άλλου είδους αποστολές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε την ειδική ε, ε, αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ. Δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις πλευρές, δεν μπορούν να επαληθεύσουν όλα όσα χρειάζεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει και ας ε, προσπαθήσουμε να στηρίξουμε προς το παρόν αυτή την αποστολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Είμαι πραγματικά ε, ε, λυπάμαι πραγματικά που χρειάστηκε να περιορίσω το χρόνο της ομιλίας. Θέλω όμως να σας ε, ε, διαβεβαιώσω ότι ο κύριος Βίγκαντ εκπροσωπεί θεσμικά όργανα και θα μπορέσουμε να τον υποδεχτούμε και άλλες φορές σε εσωτερική συζήτηση. Εάν αισθάνεστε ότι θα πρέπει να ε, επεκταθείτε σε κάποια από αυτά τα θέματα, σας παρακαλώ να υποβάλλετε γραπτές παρατηρήσεις. Εάν χρειαστεί, θα απέχω από το να ε, κάνω προφορικά συμπεράσματα, παρότι προβλέπεται από το έγγραφο. Ενδεχομένως θα έχουμε μια κοινή δήλωση η οποία είναι τώρα υπό διατύπωση για λίγη ώρα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριοι πρέσβεις και κύριοι διευθυντές που ήρθατε εδώ. Θα γίνει τώρα η δημόσια ακρόαση σχετικά με την δραστηριότητα των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας εντός του πλαισίου Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας. Σας ευχαριστώ.